Madame le Président, Bonjour à tous. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όσους είναι παρόντες. Άρχεται η Σύνοδος. Η σε διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση